Ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ είχα να κάνω την, την ανακοίνωση για τον κύριο Μπέ και την ανακοίνωση της κύρωσης κατόπιν επαλήθευσης των γεγονότων και περνάω